Ε, Η κυρία Βαλεάν ε, έρχεται σε ένα-δύο λεπτά. Η πρόεδρος της ΕΝΒΗ. Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Uh, Αγαπητοί φίλοι, περιμένουμε για να αρχίσει η συνεδρίασή μας, γιατί είναι κοινή συνεδρίαση. Γιατί οι συνάδελφοι από την Ένβη ε, πρέπει επίσης να έρθουν, μαζί με την κυρία Βαλεάν. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε χωρίς να έχουμε κανέναν από την Ένβη. Οπότε λυπάμαι, αλλά πρέπει να περιμένουμε. If we've got somebody from Envy. Είναι κανείς από την Envy. Θα ήταν καλό να έχουμε κάποιον από την Envy. Α, ωραία. Ίσως να μας συγχωρήσουν αν ξεκινήσουμε χωρίς την κυρία Συμπρόεδρο. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Έχουμε κάποια διαδικαστικά θέματα και άλλα. Πρώτα απ' όλα έγκριση μερίσιας διάταξης. Την έχετε την, κοινή, την ε, ημερήσια διάταξη για την κοινή μας συνεδρίαση. Έχετε παρατηρήσει όχι. Ωραία ανακοινώσει. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή e-meeting είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη ήτρε και ένβη τους βοηθούς και τις πολιτικές ομάδες στις ταμπλέτες ή τα λάπτοπ για να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της συνεδρίασης. Αυτό είναι καλό μια που δεν έχουμε την ε, συμπροεδρεύουσα, αλλά θα μπορεί να τα δει αργότερα. Δεύτερο, τρία μάλλον. Είναι το, ε, η έκθεση για τη διακυβέρνηση της Ελληνική Ένωσης. Είναι ο κύριος Τούρμες από την Ήτρε, από τους Πράσινους και μισό Ριβαζή από τους Πράσινους, Envy. Θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. Οι δικές μου παρατηρήσεις. Α, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ριβαζή δεν είναι εδώ. Η κυρία Ριβαζή. Ο Κλοντ βεβαίως όπως πάντα είναι εδώ. θα μπορέσει να παρουσιάσει την άποψη και των δύο εισηγητών. Διαδικαστικές παρατηρήσεις. Καλώς ορίσατε και από τις δύο επιτροπές. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία, ιδιαίτερα την κυρία Βαλεάν, η οποία είναι ακόμη εδώ, και τους δύο συνεισηγητές, τον κύριο Τούρμες και την κυρία Ριβαζή, η οποία μάλλον θα είναι την επόμενη φορά. Λοιπόν, η έκθεση θα συζητηθεί και θα εγκριθεί σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και άλλε κοινέ συνεδριάσει των δύο επιτροπών. Θα υπάρχει χωριστή ημερήσια διάταξη για κάθε μία από αυτέ τι ε, κοινέ συνεδριάσει. Να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε συμφωνήσει και οι δύο επιτροπέ ότι οι κοινέ αυτέ συνεδριάσει θα συμπροεδρεύονται από του δύο προέδρου. Το επόμενο θέμα. Προβλέπετε μια μισή ώρα για την συζήτηση αυτής της έκθεσης. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον εισηγητή μας, τον μόνο παρόντα, και μετά τους κοιόδης. Λοιπόν, να πω και δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, ενεργειακή ένωση, οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Έχουμε πολλούς στόχους και πρέπει λοιπόν να τους εφαρμόσουμε πλήρως για να έχουμε μια πραγματική και βιώσιμη ενεργειακή ένωση. Πρέπει να εφαρμόσουμε όλες μας αποφάσεις και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι το πιο σημαντικό θέμα, το κύριο θέμα για τη διακυβέρνηση της Ένωσης. Εάν δεν υπάρχει μια δομή διακυβέρνησης διαχειρίσιμη ε, που να βασίζεται στην αγορά και τις επενδύσεις και που να προστατεύει την επικουρικότητα δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η έκθεση είναι τόσο σημαντική. Γιατί είναι ακριβώς για τη διακυβέρνηση. Και μάλιστα για να βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους που περιέχονται σε άλλες εκθέσεις του πακέτου για την καθαρή ενέργεια, συνολικά οκτώ εκθέσεις όπως ξέρετε. Οκτώ νομοθετικές προτάσεις, η μία αφορά τη διακυβέρνηση. Οι στόχοι λοιπόν αναφέρονται σε 7 άλλες εκθέσεις. Χαίρομαι που οι δύο εισηγητές για την ε, οδηγία για την καθαρή ενέργεια, οι κύριοι Μπλάνκο Λόπεθ και Γκέρεκ, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι παρόν. Ευχαριστώ όμως τους παρόντες ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ welcome to all of you, colleagues from Envy Committee, each all together. I will shift your the the the floor after 20 minutes, something like that. Okay? Now I I will ask. Ο κύριος Τούρμες, ο εισηγητής μας. Να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης αλλά και την έκθεση της κυρίας Ριβαζή. Κλώτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Μισελ Ριβαζή χρειάστηκε να πάει στο γιατρό. Αλλά είναι μια χαρά. Σήμερα όμως δεν μπορούσε, γιατί έπρεπε να κάνει μια εξέταση. Διαβάσατε νομίζω την κοινή έκθεση Νομίζω ότι είναι καλή αυτή η νέα διαδικασία ότι συνεργαζόμεθα με τους συναδέλφους από την ΕΝΒΗ γιατί η κλιματική και ενεργειακή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες επί των προτάσεων μου. Νομίζω ότι διαβάσατε να επισημάνω μερικά βασικά. Χρειαζόμαστε κοινό προπολογισμό για να καταλάβουμε ότι είναι Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλές δαπάνες τώρα, αλλά στην επόμενη δεκαετία πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να φτάσουμε στο σημείο καμπής. Ο Επίτροπος Μοέντας ε, που θα είναι το απόγευμα θα μας πει ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο μηδέν και στις μεταφορές και στην ε, οικιακή χρήση και θεωρώ ότι το μηδέν θα είναι πιο εύκολο στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Το άλλο θα είναι, τα, οι άλλοι δύο τομείς θα είναι πιο δύσκολοι. Οπότε, η αλληλουχία, η χρονική αλληλουχία που προτείνει η Επιτροπή είναι πρώτα το πρόγραμμα για το 2030 και μετά από τρία χρόνια το πρόγραμμα για το 2050 δεν είναι νομίζω η καλύτερη λύση. Πρέπει παράλληλα οι κυβερνήσεις να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν πώς θα φτάσουν στο 2050 και μετά βέβαια να πούν πολύ περισσότερα για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη δεκαετία. Δεν μπορεί να διατυπωθεί ένα δεκαετές πρόγραμμα εάν δεν έχουμε υπόψη την ε, προοπτική μέχρι το 2050 και δεν θα μπορούσαν να γίνουν σωστές επενδύσεις η Ενεργειακή Ένωση, όχι μόνο η διακυβέρνηση αλλά συνολικά λοιπόν, η Ενεργειακή Ένωση θα, δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, νέα μορφή της οικονομίας μας αλλά και νέα γεωπολιτική. Κοιτάξτε τώρα τι λένε στις ε, συνεδριάσεις ε, μετόχων των ε, πετρελαϊκών εταιριών. Όλοι θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην ακμή της χρήσης της, ε, του πετρελαίου. Από τη μία λοιπόν έχουμε την ε, Ρωσία, την Αμερική και την Σοδική Αραγία που παράγουν πετρέλαιο και από την άλλη μεριά η Ευρώπη, η Ινδία και η Κίνα είναι αυτοί που είναι πρωτοπόροι τεχνολογία και στο μέλλον ε, η ευημερία θα είναι σε αυτούς που έχουν περισσότερη τεχνολογία. Εμείς έχουμε τόσο καλό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε τόσο καινοτόμες εταιρείε. Είμαστε πρωτοπόροι τεχνολογία. Έχουμε λοιπόν λαμπρό μέλλον, αλλά θα το επιτύχουμε μόνο αν δράσουμε από κοινού. Το σύνθημά μου λοιπόν είναι ότι οι κυβερνήσει πρέπει να δράσουν από κοινού μαζί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα καλό πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των πολιτών. Και για όλα αυτά, αυτό που χρειάζεται είναι και εμείς ως πολίτες και οι κυβερνήσει να πιστούν ότι, ότι απέχουμε ακόμη πολύ από την ε, ευαισθητοποίηση των πολιτών. Βεβαίως μπορούμε να πείσουμε τους φορείς που συμμετέχουν, αλλά νομίζω πως θα ήταν ε, αλαζονία να θεωρούμε ότι εμείς από τις Βρυξέλλες ή από το Βερολίνο μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Όχι, πολύ πιο κοντά είναι ο Δήμαρχος της Κοπενχάγης ενός χωριού. Αυτοί θα μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν. Γι' αυτό νομίζω ότι η προσέγγιση της Επιτροπής ε, είναι παραδοσιακή. Θα ενημερώσουμε για την κοινή γνώμη. Όχι, όχι. Πρέπει να τους κινητοποιήσουμε σε στρατηγική συνεργασία με τις πόλεις. Και αυτό θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας και στην Ήπεθρο. Η, ε, τα αιωλικά πάρκα δεν είναι στο κέντρο των πόλεων, είναι στην Ήπεθρο. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ερημώνει η Ήπεθρός μας. Και αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν έτσι να έρθουμε σε επαφή με την Ήπεθρο, τους κοινοτάρχες κτλ. Και μετά βέβαια πρέπει να ασχοληθούμε και με τις επενδύσεις. Δεν θα αρκέσουν οι δημόσιες. Πρέπει να υπάρξουν και ιδιωτικέ. Και αν θέλουμε ιδιωτικέ επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα. Ένας επενδυτής πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ε, μηδενικές εκπομπές ε, ορυκτών καυσίμων το 2050 και αμέσω τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Τι απόδοση θα έχει η επένδυση μου. Αυτό χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι εάν έχουμε καλά σχεδιασμένε αγορέ και ε, απευθύνομαι στου συναδέλφου από το ΕΛΚ, τον Κούναρ και τον Κρίστιαν, νομίζω ότι το ΕΛΚ θα μα βοηθήσει για να σχεδιάσουμε καλύτερα τι αγορέ, αλλά θα υπάρχει και ένα τμήμα προγραμματισμού γιατί για να ξεκινήσει η ηλεκτρική κινητικότητα χρειάζεται να έχουμε ε, σημεία φόρτισης. Η, η τηλεθέρμανση χρειάζεται προγραμματισμό, χρειάζεται σχέδια, χρειάζεται η δυνατότητα των θεσμών στις πόλεις και τα χωριά των θεσμικών οργάνων. Βλέπω την Κεζίνε Μάισνερ. Αν θέλουμε οι κυβερνήσεις να έχουν ε, την ε, πρωτοβουλία για να αναπτύξουν ανεμογεννήτριες υπερακτίως, χρειάζεται οι κυβερνήσει να κάνουν το σωστό προγραμματισμό. Ο προγραμματισμό, η σχεδιασμένη οικονομία δηλαδή χρειάζεται σε έναν βαθμό και άμα γίνει σωστά βοηθάει του επενδυτέ. Και τελευταίο. Πρέπει να γίνουν σωστά οι επενδύσει ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δηλαδή ο συνδυασμό των δικτύων τώρα βοηθάει τι βαλτικέ χώρε να εξαρτώνται λιγότερο από τη Ρωσία που θα βοηθήσει να συνδεθούν η Γαλλία με την Ισπανία, που θα βοηθήσουν η Ιρλανδία να συνδεθεί με την υπηρετική ε, Ευρώπη αν η Βρετανία ε, πλεύσει προς το Τέξας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την ενεργειακή φτώχεια στην Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ευφυή σχεδιασμό για ευφυή κτίρια. Χρειαζόμαστε λοιπόν επαρκείς πιστώσεις για ανανεώσιμες, για υπεράκτη αιωλικά πάρκα, να μειωθεί το κόστος, ε, το κόστος των επενδύσεων στη Ρουμανία, την Πολωνία, την Βουλγαρία. Γιατί να μην υπάρχει δυνατότητα και ακόμη και πολίτες να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις εάν αποφασίσουν, για παράδειγμα, να στήσουν ανεμογεννήτριες και χρειάζονται κάποια βοήθεια, κάποια επιδότηση για κάποια χρόνια. Πρέπει λοιπόν περισσότερο και στην περιφερειακή πολιτική να ρεύσουν περισσότερο απευθείας πιστώσεις για να κινητοποιηθούν περισσότερο. Να αποδεσμεύσουμε, να απελευθερώσουμε τη μεγάλη μας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχατε 10 λεπτά για δύο εισηγητές, αλλά εσείς ήσασταν πιο σύντομος. Σκιώδης τώρα του ΕΛΚ η κυρία Ντελαέ, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ο κύριος Χόκμαρκ από την Ήτρη. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι δεδομένη της καθυστέρησης και των υποχρεώσεών μου δεν μπορώ να μείνω μέχρι το τέλος της συζήτησης αλλά επειδή συνεργάζομαι πολύ στενά με τον συνάδελφο θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε τα όσα θα υποθούν σε διάρκεια αυτής εδώ της Μικτής Επιτροπής συνεδρίαση μάλλον των επιτροπών μας, ε, Ενβι και Εγώ κατάλαβα πολύ καλά τα όσα μας είπε ο συνάδελφος ε, για τα περιβαλλοντικά διακυβεύματα αλλά και τα στρατηγικά διακυβεύματα. Εγώ είμαι, κάποιος, ε, είμαι πολύ ρεαλίστρια, προέρχομαι, είμαι από την πολύ κοντά στη γη και γνωρίζω τα όσα λέγονται για την ενέργεια και τη διακυβέρνηση αυτής, ότι δηλαδή αυτή η διακυβέρνηση πάνω απ' όλα είναι μια ενότητα η οποία θα καλύψει το σύνολο των οδηγιών που αφορούν τα ενεργειακά θέματα. Και έτσι για να συμβαστούμε και τη συμφωνία, του, τη συμφωνία των Παρισίων θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται πάνω απ' όλα για ένα εργαλείο συντονισμού ε, σε θέματα συνεργασίας περιβαλλοντικής και κλίματος. Ε, θα πρέπει να μην είμαστε ιδιαίτερα περιοριστικοί και ορισμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Για να έχουμε έναν κατάλογο μέτρων θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν στις οδηγίες καλύτερα ε, και ακριβώς εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε και για τους στόχους όσον αφορά τις ανανεώσιμες, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και όχι μέσα στην ε, γενικότερη ε, ε, ομπρέλα που εδώ καλούμεθα να φτιάξουμε. Θέλω να μιλήσω λίγο για τη μέθοδο, γιατί ακριβώς οι μέθοδοι είναι αυτές ε, οι οποίες είναι διαφορετικές, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά προβλήματα να αντιμετωπίσει σε σχέση με την ενέργεια και το κλίμα. Γι' αυτό θα πρέπει συλλογικά να δούμε τι θα κάνουμε, ώστε συλλογικά να πετύχουμε ε, στην ευρωπαϊκού στόχους τους οποίους έχουμε θέσει και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, θα πρέπει να επιτρέψουμε μια κάποια ευελιξία, να λάβουμε υπόψη το οικονομικό περιβάλλον κάθε κράτους μέλους, γιατί τα πράγματα διαφέρουν από τη Δύση στην Ανατολή και από το Βορρά στο Νότο της Ευρώπης, αλλά πρέπει από κοινού να επιδιώξουμε αυτόν τον κοινό στόχο που έχουμε θέσει. Έχω μια παρατήρηση επί του ουσία τώρα όσον αφορά το ETS, γιατί αυτήν ε, αντιμετωπίζεται στα παρατήματα και όχι στο διατακτικό του κειμένου. Δεδομένου αυτού όμως του θέματος και των συζητήσεων που κάνουμε, πιστεύω πως το ETS θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του διατακτικού και να κλείσω λέγοντα ότι αν, μείνουμε, αν είμαστε ρεαλιστές και αν επιτρέψουμε στον καθένα να εξελιχθεί ανάλογα με την κατάστασή του, περιορίζοντα τον, ε, δημοσιο... τον ε, διοικητικό φόρτο, μην ξεχνάμε ότι αυτή η θητεία είναι υπό την αιγίδα τη καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να σκεφτούμε και τι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, την πρόοδο τεχνολογική που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς μας στόχους και ότι θα πρέπει περισσότερο να εθαρρύνουμε, αντί να θέτουμε βερβολικά φιλόδοξους στόχους, πολύ γρήγορους και πολύ απομακρυσμένους, να ακολουθήσουμε από κοινού την ίδια κατεύθυνση για την επίτευξη αυτό. και πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι το καλύτερο είναι ο εχθρό του καλού πάντα. Ο συνάδελφος Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους εισηγητές και την Σκιώδη συνάδελφο. Εγώ θέλω να προσθέσω κάποιες σκέψεις. Η πρώτη είναι αυτή που ανέφερε ο κύριος Τούρμες, ότι δεν χρειάζεται, ε, το, όταν μιλάμε για σχεδιασμό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε κομμουνιστές. Συμφωνώ με αυτό. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν θα πρέπει τα σχέδια να πάρουν μεγαλύτερη σημασία από την πραγματικότητα, γιατί τότε θα έχουμε προβλήματα. Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο χάρτη και την πραγματικότητα, καλύτερα είναι να ακολουθήσουμε την πραγματικότητα. Έτσι λέει ένα ρητό. Και αυτό είναι το, αυτή είναι η ισορροπία που θα πρέπει εμείς να διατηρήσουμε. Γιατί κατά τη γνώμη μου ε, το σημαντικό δεν είναι ο αριθμός των στόχων, δεν είναι ο αριθμός των εκθέσεων, ούτε ο αριθμός και το μέγεθος των σχεδίων μας. Είναι ο μηχανισμός και οι δομές που θα φτιάξουμε, που θα μπορέσουν να μετατρέψουν σε πραγματικότητα την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και με την Ενεργειακή Ένωση, αν αυτή λειτουργήσει εύρυθμα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. και για το στόχο του κλίματος και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα προκύψουν από την εξέλιξη και την, την ανάπτυξη αγοράς, όχι από τις επιδοτήσεις και τα σχέδια. Θα προέλθουν από τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την ανοιχτή αγορά. Και γι' αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τις δομές ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την ε, Ε, συνεργασία όχι από πάνω προς τα κάτω αλλά να διευκολύνουμε το διασυνοριακό εμπόριο, διαμεθοριακό εμπόριο ε, να στηρίξουμε τις διασυνδέσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε όλες τις ε, πηγές ενέργειας και γι' αυτό και χρειάζεται να είμαστε προσανατολισμένοι στην αγορά γιατί διαφορετικά θα έχουμε τελματωμένες δομές. Να εξασφαλίσουμε ότι το ενεργειακό μείγμα θα εξαρτάται από τα κράτη-μέλη αλλά ότι πρέπει ωστόσο να συνεργαστούμε πολλά από τα πράγματα που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμή σήμερα, αλλά και τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε ε, στην έκθεση, μας δίνουν τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Πιστεύω ότι στον βασικό τομέα έχουμε πάνω κάτω τους ίδιους στόχους. Η διαφορά μας είναι το πώς αυτούς θα τους πετύχουμε. Εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε προτεραιότητα στο να εξασφαλίσουμε το ότι στην πραγματικότητα προχωρούν στη σωστή κατεύθυνση τα βήματά μας μέσω του διαμεθοριακού εμπορίου, του, της ανοιχτής αγοράς, των νέων τεχνολογιών. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση και βεβαίως προσβλέπουμε στις συζητήσεις μαζί σας. ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους και από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο κύριος Σοχίνιο. Ή μήπως ονειρεύομαι. Ε, από την Εύη ή την Ήτρε. Όχι. Τώρα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Εύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση αυτή έχει θεμελιώδη σημασία και θα καταστήσει πιο διαφανή την πολιτική διαδικασία λήψη απόφαση ε, στην Ενεργειακή Ένωση. Και θα ήθελα να συγχαρώ τους συγητές ε, για την καταπληκτική τους προσπάθεια και τη φιλοδοξία τους να ευθυγραμμίσει τις ενεργειακές πολιτικές με τη Συμφωνία των, Παρισίων. Ε, άσκησα το ρόλο του Σκιώδου του στην ΕΜΒΗ ε, με αγαστή συνεργασία, σε αγαστή συνεργασία με την Τερέζα Γκρίφιν, την σκιώδη συγκήτρια από την Ήτρε. Και από κοινού θα συντάξουμε μια σειρά τροπολογιών για να συμπληρώσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ενισχύσουμε κάποιες από τις ιδέες της έκθεσης. Εν συντομία, για να συμπληρώσω αυτό που θα πω αργότερα και η Τερέζα, γιατί είναι κοινέ οι προτάσεις μας, η πρώτη μας ιδέα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συνεισφέρουν μόνο στην πολιτική. Θα πρέπει να υπομισθούν και κάποιες ευθύνες. Γι' αυτό και προτείνουμε δεσμευτικούς στόχους. Οι δεσμευτικοί στόχοι θα πρέπει να εθιγραμμίζονται με τους στόχους σε άλλα θέματα. 35% για τις ΑΠΕ, για την ενεργειακή απόδοση, 40%. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση των στόχων. Αυτό έχει νόημα, η συνοχή. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης, ε, τα σχέδια ενέργειας και κλίματος για το 2003 θα πρέπει να συνδέονται με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές και πέραν του γνώμονα του Γενικού Υποδείγματος για το 2030 θα πρέπει να έχουμε και υποδείγματα για μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να εξασφαλίσουμε μια συγκρισιμότητα μεταξύ αυτών των στρατηγικών. Επίσης, ε, προτείνουμε πενταετή σχέδια ενεργειακά για να θυγραμμίσουμε τα τους προθεσμίες της διακυβέρνησης με τις προθεσμίες που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Όλα αυτά έχουν νόημα όταν είναι αναπόσπαστα τμήματα ενός συνόλου. Επίσης θα προτείνουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην διαμόρφωση των σχεδίων, μεγαλύτερη διαφάνεια των σχεδίων και επίσης προτείνουμε τη σύσταση ενός δίκαιου ταμείου ε, μεταβασής ε, ώστε να διευκολύνουμε αυτή την μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Θα προτείνουμε τροπολογίες για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις κάποιων πολιτικών. Θα ταχθούμε υπέρ της περιφερειακής ολοκλήρωσης ε, των χωρών και συμβασμό τους με, τις, με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Τερέζα που είναι μεγάλος υπέρμαχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και έκανε ως λάβαρό της την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτές οι γενικές γραμμές είναι η πρότασή μας και σίγουρα η συνάδελφος η Τερέζα Γκρίφιν, η σκιώδη συνεισηγήτρια, θα συμπληρώσει τα δικά μου σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκρίφιν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γέζη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ευχαρισ... τις ευχαριστίες μου προς τον Κλοντ για την αγαστή συνεργασία ε, των δύο επιτροπών Ιτρεκέμβη. Όπως είπε και ο Κάρλος, ε, ε, η πρόταση των συνεισηγητών βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ήταν μέχρι στιγμής εξαιρετική συνεργασία. Αυτό που επιδιώκουν οι συνεισηγητές είναι να μεταστρέψουν από την έκθεση από μία απλή ε, έκθεση για την ενεργειακή διακυβέρνηση σε μία γενικότερη πολιτική που υπό το πρίσμα του κλίματος και της ενέργειας θα παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές. Συμφωνώ και επίσης είμαι υπέρ της ευθυγράμμισης των εθνικών ε, σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας. Έτσι θα καταφέρουμε ε, τους φιλόδοξους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων να τους συμπεριλάβουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όπως είπε ο Κάρλος, θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τους κανονισμούς σε εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για τις ανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την, την συμμετοχή των ενδιαφερομένων και στην χάραξη, ανάπτυξη αλλά και στην εφαρμογή των σχεδίων και θα πρέπει τα σχέδια και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας να είναι διαφανή για να το καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Επίσης, Είμαστε υπέρ μια διασυνοριακή στρατηγική και για τα σχέδια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, όπω είπε ο Κλοντ. Ω και όδη ηγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θα ήθελα να υποβάλω τροπολογίε προκειμένου να ενισχύσουμε το κείμενο σε δύο τομεί. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή φτώχεια, θα πρότεινα τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν την έννοια της ενεργειακής φτώχειας και το, την έννοια των ευάλωτων καταναλωτών με βάση δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορούν να συγκεντρώνουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα στα πλαίσια του νέου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Ένδυα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα κράτη-μέλη μπορούν να θέσουν ως στόχο να μειώσουν τον αριθμό των ευάλωτων καταναλωτών και να ευθυγραμμίσουν τα ενεργειακά του σχέδια με το στόχο αυτό της καταπολέμησης ενεργειακής ένδυας. Επίσης, όπως είπε ο Κάρλος, είμαι υπέρ της α, υιοθέτηση μιας πρωτοβουλίας για δίκαιη μετάβαση. Γιατί μια ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα σε εργαζόμενους και ορισμένε περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μια τέτοια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δίκαιη μετάβαση θα στηρίξει αυτούς τους πολίτες ώστε να κάνουν και αυτή τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Θα χρηματοδοτεί κοινοτικά σχέδια για επανακατάρτιση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων ε, των εργαζομένων, προκειμένου να κάνουν πιο ομαλά τη μετάβαση και θα στηρίξει και νέες υποδομές. Επαναλαμβάνω, θα συνεργαστούμε επικοδομητικά, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και τις πόλεις, προκειμένου να φέρουμε τους πολίτες στο επίκεντρο αυτής της Ενεργειακής Ένωσης. Ευχαριστώ. ECR τώρα. Ο εκπρόσωπο του ECR για την ΕΜΒΗ δεν είναι παρόν. Ο συνάδελφο του Ζενόφσκι. Που μιλάει εκ ονόματο και των δυο εισηγητών. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γιάζη. Eh, Σας ευχαριστώ. Eh, Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την πρόταση και θέλω να ευχαριστήσω και για τη δυνατότητα που μας δώσατε να συζητήσουμε με τόσο λεπτομερή τρόπο αυτή την έκθεση που είναι τόσο μεγάλη σημασία. για μια έκθεση που θα πρέπει να την ψηφίσουμε με στη διάρκεια αυτού του έτους. Οπότε η συνεργασία μεταξύ των εισηγητών και των σχεδόν εισηγητών είναι πολύ σημαντική. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τη νομοθετική διαδικασία και να την απαλλάξουμε από περιτέ ε, περιπλοκές. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των εθνικών σχεδίων που οφείλουν να είναι αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να γίνουν αντιληπτά στο ευρύ κοινό, στους πληθυσμούς των χωρών μελών. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ιδιαίτερα διεξοδική. Περιλαμβάνει όμως ε, περιττό διοικητικό φόρτο ε, για την προετοιμασία τέτοιων σχεδίων. Οπότε οι προτινόμενες απλουστεύσεις είναι πολυδόκιμες. Χρειάζεται κάποια απλοποίηση εδώ για να περιορίσουμε το διοικητικό φόρτο και δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο διεξοδικοί ως προς λεπτομέρειες. Έχω όμως ένα πρόβλημα και η ομάδα μου δεν συμφωνεί με κάποια σημεία και κυρίως με τους στόχους του εισηγητού, όπως τους παρουσιάζει στην πρόταση. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι στο με αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε ενιαίους στόχους, γιατί οι στόχοι συνδέονται και με άλλους παράγοντες και πτυχές και αν έχουμε ενιαίους δεσμευτικούς στόχους θα υπάρξει πρόβλημα. Και θα δημιουργήσει η υπάρξη τέτοιων ενιαίων στόχων υπερβολικές επιπλοκές στα κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνω, η πρόταση δεν θα πρέπει να είναι περίπλοκη. Θα πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις εθνικές τους πολιτικές προσαρμόζοντάς τις τις ανάγκες τους. Εμείς έχουμε πρόβλημα με τον οριζόντιο, αυτό το γραμμικό παράγοντα που επηρεάζει τον οικονομικό κύκλο και άλλες ε, επιμέρους ε, ρυθμίσεις. Κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτη η θέσπιση νέων στόχων. Αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει εμείς να επιβάλλουμε νέους στόχους. Επίσης, αυτό το 40% που προτείνουμε ως στόχο για την ενεργειακή απόδοση δεν στηρίζεται σε επιστημονικά πορίσματα και πολλές χώρες αφισβητούν αυτό το στόχο και θα καταφέρουν να να τον υλοποιήσουν. Επίσης μιλάμε για το 30% των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Για πολλές χώρε και αυτός ο στόχος είναι δυσβάσταχτος. Θα καταφέρω λοιπόν πολλές χώρε να ε, υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό και η ομάδα μου έχει σοβαρές αμφιβολίες και ως προς το ενεργειακό μείγμα. Η σύνθεση του ενεργειακού μείγματος είναι εθνική αρμοδιότητα. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση δεν εξασφαλίζει την επαρκή διακριτική ευχέρεια και ελευθερία λήψη αποφάσεων στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ενεργειακού του μείγματος. Ε, ε, νομίζω ότι επιβάλλει πολλά πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι για τη συνεργασία. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν πολλέ συζητήσει και ελπίζω να καταφέρουμε από κοινού να καταλήξουμε σε κοινέ προτάσει, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και θα είναι σημαντικά και στο μέλλον θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που καλύψατε τα σχόλια και των δύο ε, εισηγητών του ECR. Εξαντλήσατε το εξάλεπτο. Παρόμοια κατάσταση έχουμε και στους φιλελεύθερους. Ο κύριος Γκερμπράντι, εκπρόσωπος της ΕΜΒΗ, απουσιάζει, οπότε η... Αλλά και η Καρολίνα από η και τη σύντρια, απουσιάζει. Η κυρία όμως Μάισνερ, που είναι παρούσα, θα καλύψει και τους δύο συνεισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εξαντλήσω κάτω εξάλεπτο, οπότε θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και νωρίτερα τη συνεδρίασή μας. Όπως είπατε, ο κύριος Κερμπράν της ΕΜΒ και η κυρία Σπόσερ της ε, Ήτρε απουσιάζουν και οι δύο και εγώ θα τους αντικαταστήσω επισημένοντας τα εξή. Καταρχήν, να χαιρετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει πολλά θετικά σημεία όπως είναι η δεσμευτική στόχη και κάτι που θα εξασφαλίσει συγκρισιμότητα και θα απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά του σχέδια με τις πορείες του 2021 και 2030 σε ό,τι αφορά τις εθνικές συνεισφορές για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση. Είναι σκόπιμο να έχουμε δεσμευτικούς στόχους για να απαιτήσουμε λογοδοσία από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, χρειαζόμαστε και μια ισχυρή διακυβέρνηση για να ε, επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Ε, για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου για του επενδυτέ, Οπότε θέλουμε και συγκριτικού κανόνε ε, με σαφεί διατάξει για τη συνεισφορά των κρατών μελών στον χρηματοοικονομικό μηχανισμό. Και από την άποψη ασφάλεια δικαίου για του επενδυτέ, τονίζουμε τη σημασία που έχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική που υπερβαίνει τον ορίζοντα του 2030. Κάτι τέτοιο είναι ζωτική σημασία για να αποδεσμεύσουμε ε, επενδύσει κυρίω για μείζονες υποδομέ με μεγάλη διάρκεια ζωή. Η υποχρεωτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων επίσης είναι θετικό σημείο και θα θέλαμε να την ενισχύσουμε. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε και στα εθνικά σχέδια να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ήδη από τη χάραξη, ε, αλλά και την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων κλίματος και ενέργειας. Θα καταθέσουμε λοιπόν σχετικές τροπολογίες και προσβλέπουμε σε καρποφόρο συνεργασία με τους δύο συνεισηγητές και τους υπόλοιπους σκιώδης συγητές. Αυτά από τους σκιώδης συγητές μας, αλλά να κάνω και κάποια προσωπικά σχόλια, να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τον πολύ ενθουσιώδη και παθιασμένο τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε την έκθεση που ακολουθεί πολλά σωστά σημεία και εκθε, ε, ε, κατευθύνσεις. Συμφωνώ με τη στρατηγική συνεργασία που επισημάνατε για τις πόλεις. Μην ξεχνάτε όμως και τις αγροτικές περιοχές, ε, την Ήπεθρο. Θα πρέπει και αυτή να, να την εμπλέξουμε στην συνεργασία. Επίσης αναφερθήκατε στο συνδέοντο στην Ευρώπη για τα δίκτυα. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και το συνδέοντα στην Ευρώπη το συνδέσαμε με τις μεταφορές ε, και τις ε, ΑΠΕ, τις ανανάσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν ε, τα δίκτυα και στις υποδομές για την ενέργεια. Γιατί είναι απαραίτητο, γιατί θέλουμε ο ήλιος που ήταν κυρίως στο νότο τώρα είναι παντού να αξιοποιήσουμε τον ήλιο από τον νότο και τον αέρα από το βορρά παρόλο που έχουμε ολική ενέργεια και στο νότο να το συνδυάσουμε ή ακόμη και την μελλοντική ενέργεια που θα μπορούμε να, να χρησιμοποιήσουμε από, το, από τα κύματα, από τους ωκεανούς, ώστε να συνδυάσουμε το δυναμικό, το αιωλικό, το ηλιακό από τις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή και γι' αυτό χρειαζόμαστε τα δίκτυα. Και θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές στη Γερμανία ε, δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος και δεν αξιοποιούνται τα δίκτυα γιατί ο, ο κόσμος θέλει να έχει τον κήπο του, αλλά αν πείσουμε τους πολίτες ότι χρειαζόμαστε για την Ενεργειακή Ένωση τα δίκτυα και θα πρέπει να δώσουμε μάχη για μια ε, αποτελεσματική ενεργειακή ένωση παντού, ίσως έτσι πείσουμε τον κόσμο να στενιστεί αυτό το σχέδιο και να προσφέρει περισσότερο στα δίκτυα. Ευχαριστώ θερμά και πιστεύω ακράδοντα ότι θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας και κάποια στιγμή θα υλοποιήσουμε, ελπίζω στο εγγύς μέλλον, την ενεργειακή μας ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, για τις παρατηρήσεις σας και ο συνάδελφος Ζωάου Φερέιρα. Από την Ήτρε δεν είναι παρόν, αλλά η συνάδελφος Καταζίνα Κονέτσινα της ΕΝΒΗ είναι επίσης κοιόδης εισηγήτρια, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ μπορείτε να μιλήσετε εξ ονόματος και των δυο σκιωδών. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ούτως οι ε, απόψεις μας είναι παραπλήσει, αλλά θα μιλήσω βεβαίως ε, από πλευράς του εαυτού το Νοέμβριο του 2016 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά νομοθετικών προτάσεων καθαρή ενέργεια για όλους και ενεργειακή ένωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ο τίτλος. Είναι βασικό κείμενο για την εφαρμογή για να επιτύχουμε τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης που είναι στα πλαίσια της πολιτικής μας για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2030. Γιατί λοιπόν το έγγραφο αυτό είναι το πρώτο που συζητάμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κοιτάξτε τι σοβαρό πρόβλημα έχουμε με το κλείσιμο του προηγούμενου πακέτου, το οποίο το έχει και το Συμβούλιο. έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα γιατί θεωρήθηκε ότι παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Δεν το καταλαβαίνουν τι οι αγορές. Δεν είναι δυνατόν επίσης να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως διάφορες προτάσεις όπως θα ήταν αναγκαίο. δηλαδή η προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2018 εξαρτάται και από τις ε, διαπραγματεύσεις για ε, το ETS. Αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου υπήρξαν έξι συνεδριάσεις ε, των, έχουν προγραμματιστεί 7 ή 8 συνεδριάσεις στο σκιωδών, αλλά δεν θα κλείσουμε το ETS. Αυτό θα γίνει από την επόμενη Προεδρία και το ESR θα, ε, θα το συζητήσουμε τον Οκτώβριο και το Λούλου CF ούτε καν ξέρουμε πότε. Δηλαδή, έχουμε μεν μία μέθοδο, αλλά όλα αυτά τα θέματα δεν γνωρίζουμε πώς θα προωθηθούν. Δεν είναι δυνατόν να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί να εγκρίνουμε για ορισμένα θέματα ένα, με βάση ορισμένα δεδομένα που δεν θα για άλλα. Στην ουσία είναι ένα παιχνίδι που γίνεται αυτό. Όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερως καλά επεξεργασμένα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η προσπάθεια. Από τη μία μεριά μας λέτε ότι έτσι θα μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων που χρησιμοποιούν άνθρακα. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Στην ουσία η μείωση της κατανάλωσης θα οδηγήσει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Αυτό που δεν έχουμε είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κύριο μέσο ε, μείωσης του άνθρακα. Οι ανανεώσιμες μέχρι στιγμής δεν έχουν προωθηθεί αρκετά. Άρα, συνολικά δεν είναι πολύ αποτελεσματικό αυτό το μέσο. Η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω δηλειτουργίες. Όμως όλα αυτά δεν αναφέρονται στην έκθεση. Πρέπει να καταλάβουμε σαφώς και να έχουμε συνείδηση ότι εδώ είμαστε Επιτροπή Ήτρε και πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι στην ενέργεια όλα συνδέονται και αν δεν λειτουργεί ένα στοιχείο της προσπάθειας καταραίει το σύστημα. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σαφές ακόμη αυτό από όλους τους συζητητές των θεμάτων ενέργειας. Ακόμη και το Συμβούλιο δεν πιέσει. Και δεν έχουμε ιδέα πότε θα ασχοληθούμε τα θέματα αυτά. Το προσωπικό μας και η νομική υπηρεσία ασχολούνται με κείμενα τα οποία είναι εντελώς αποσπασματικά και μερικά. Γι' αυτό δεν στηρίζω να, την προσπάθεια να προωθήσουμε το θέμα αυτό τον Σεπτέμβριο θα ήταν ανεύθυνο. Γι' αυτό προτείνω την αναβολή της εξέτασης. Αλλιώς θα είναι βιβλιασμένη η προσέγγιση και η έκθεση που μας έχει υποβάλει δεν λύνει κανένα θέμα. Είναι επικίνδυνα ε, αποσπασματικά μέτρα αυτό θα προκαλέσει ζημιά στην αξιοπιστία της Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έξι λεπτά για τους δύο σκιώδεις. Για το EFDD. Ο συνάδελφος Ταμπουράνο δεν είναι παρόν. Αλλά έχουμε τον συνάδελφο Πεντιτσίνη από την Ένβη. Ε, θα μπορούσε να εκπροσωπήσει και τους δύο εκπροσώπους. Μάλιστα. Εγώ λέω πως η θέση μας η δική μου δηλαδή και του κύριου Ταμπουράνο είναι η ίδια. Έχουμε την τύχη να έχουμε κοινή γνώμη τόσο εδώ, στην, ε, μάλλον τόσο στην ΕΒ όσο και στην Ήτρε για αυτά τα θέματα. Για μας η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης σημαίνει καταρχάς υποχρεώσεις των κρατών μελών. Άρα λοιπόν πρώτα απ' όλα οι στόχοι θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί για κάθε κράτος μέλος και όχι να εξαρτώνται από την καλή θέληση καθενός. κάθε κράτος πρέπει να αναλάβει ε, την ευθύνη για την επίδειξη αυτών των στόχων. Έπειτα θα πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικό και σοβαρό σχέδιο για, ε, για κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα. Και αυτό θα έπρεπε να είναι κοινό για όλα τα κρατημέλη, εφόσον θέλουμε πραγματικά μετάβαση προ Ενεργειακή Ένωση που θα βασίζεται στι ανανεώσιμε. Η κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα για μα είναι ο μοναδικό ε, δρόμο. Ελπίζω να μην λάβουμε τις συνήθεις απαντήσεις ότι τα κατημέλη μπορούν να διαλέξουν το ενεργειακό μίξ, γιατί κατά τη γνώμη μας αυτό είναι πια γελίο. Να προσθέσω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά που έχει κάνει ο συνάδελφος Τούρμς και η συνάδελφος Ριβαζή, καθώς και, και επειδή θέλουν να ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες, ε, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Πιστεύουμε ότι τα κρατημέλη οφείλουν να είναι, μάλλον θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένα να λάβουν αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την γνώμη των ε, πληθυσμών και των τοπικών πληθυσμών, αντί να επιβάλλουν, όπως συχνά συμβαίνει, το, στις τοπικούς πληθυσμούς αποφάσεις ενεργειακού τύπου που ε, πλουτίζουν λίγους, ενώ ε, τελικά το κόστος πληρώνεται από, ολόκλη, από τους πολίτες συνολικά. Ε, Επίση, ε, θέλουμε την ε, αξιολόγηση για τις εκπομπές μεθανίου με στόχο την λήψη μέτρων για την μείωση αυτών των εκπομπών. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν κατ' τα σχόλιά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, για αυτές σας τις παρατηρήσεις. Ο κύριος Ζανλουκ Σαφχάουζερ από την Ήτρε δεν είναι εδώ αλλά είναι εδώ η κυρία Ντονανό από την Επιτροπή ΕΝΒΗ που εκπροσωπεί το ΕΝΕΦ e και μπορείτε να μιλήσετε και εξονόματος των δύο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους συνεισηγητές για την εργασία τους. Δεν μπορώ βεβαίως παρά να στηρίξω τις απαιτήσεις ε, ε, εποπτείας, παρακολούθησης, εκθέσεων και επαλήθευσης ε, με βάση την τη σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο, η Συμφωνία των Παρισίων 12 Δεκεμβρίου 2015 μας υποχρεώνει να είμαστε ρεαλιστές. Η μόνη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει την δράση διεθνών οργανισμών μεταξύ, οποίου ε, στους οποίους είναι ακόμα μέλη η ΕΠΑ σε σχέση με τους στόχους που, που ανανεώσατε για ένα ποσοστό σημαντικό για τις ανανεώσιμες το 2050 θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να αναθεωρήσουμε τους ορισμούς περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Επίσης θα πρέπει περίπτωση να αξιολογήσουμε, την κάθε περίπτωση να αξιολογήσουμε χωριστά και έπειτα θα είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Τα αιωλικά πάρκα και η βιωσιμότητά τους είναι αμφισβητήσιμη. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι αιωλικές ε, γεννήτριες έχουν ένα πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος για την κατασκευή και για τη διάλυσή τους και ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι βιώσιμα. Επίσης αυτή η πηγή ενέργειας είναι διακοπτόμενη, ε, μπορεί να κάνει ε, παράσιτα στις ε, διάφορα, σε διάφορα μαγνητικά κύματα, τηλεοπτικά και τέτοιου τύπου, καθώς και βλάπτει τους ε, πληθυσμούς πτηνών καθώς και θαλασσίων θηλαστικών Πράγμα το οποίο κοστίζει πολύ πολύ ακριβά. Ε, το ίδιο και οι, τα φωτοβολταϊκά κέντρα επίσης έχουν πολύ μεγάλο κόστος, δεν είναι πολύ δε, οικολογικά τα συστατικά, ε, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και έτσι εγκρίνω την ε, βούληση να ε, περιοριστούν οι εκπομπές μεθανίου, καθώς αυτό το αέριο είναι πολύ πιο ισχυρό όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου από ότι το ε, διοξίδιο του άνθρακα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει όλα αυτά να έχουν επιπτώσεις στους δικούς μας θυνοτρόφους ε, γιατί Εάν και, και ακόμα και αν ε, συμβάλλουν στην εκπομπή μεθανίου θα πρέπει να προστατευθούν, γιατί είναι ήδη ευάλωτοι. Θα υποβάλω τροπολογίες επικοδομητικού τύπου που ωστόσο θα είναι πάντοτε ε, σαφέστατες γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά κυρία Ντορνονό τις παρατηρήσεις. Ακούσαμε τους και ηγητές. αλλά έχουμε σκιώδεις ηγητές ε, και από άλλες εκθέσεις, για άλλες εκθέσεις και ένα κατάλογο ομιλητών. Θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο, την κυρία Βαλεάν, για να συντονίσει τη συζήτηση. Θα ήθελα... Μια και έχει ξεκινήσει η συζήτηση, να μην σταθώ σε ανακοινώσει, αλλά να συνεχίσουμε. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπούζεκ, στο πακέτο αυτό έχουμε και άλλες εκθέσεις ε, αλληλένδετες με τη συγκεκριμένη. Γι' αυτό και οι συγκητές ε, για την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να λάβουν το λόγο. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπλάνκο Λόπες, που είναι επιφορτισμένος με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Τούρμες και την κυρία Ριβαζή για το έργο τους. Θα ήθελα όμως ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε κάποια σχόλια που άκουσα. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές. Η απαλλαγή όμως της οικονομίας από τις αθρακούχες εκπομπές δεν είναι πια επιλογή, είναι υποχρέωσή μας. Και γι' αυτό χαιρετίζω την έκθεση που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του Παρισιού της COP21 και επίσης συμπληρωματική ως προς τη δική μου πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σχετική οδηγία, την αναθεώρηση τη οποίας θα συζητήσουμε αύριο. Είναι συμπληρωματικές λοιπόν οι δύο εκθέσεις και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Κάτι που προποθέτει δεσμευτικού εθνικού στόχου για κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν με συγκεκριμένου στόχου. Αυτό έχει λειτουργήσει καλά μέχρι ε, στην ε, υπάρχουσα οδηγία που προσφέρει ασφάλεια στους επενδυτές, βεβαιότητα, δέσμευση και ευκολία σχεδιασμού χάρη αυτή την ασφάλεια δικαίου. Άλλωστε έτσι θα, θα γίνει και πιο φθηνή χρηματοδότηση στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, στην καινοτομία και θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τον γενικό μας στόχο. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην πρόταση που θα σας παρουσιάσω αύριο θα υποστηρίξω 35% τουλάχιστον μερίδιο στις ΑΠΕ για το 2030. Κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό, αποδοτικό και έχει πολλά ωφέλη που ξεπερνούν τα ενεργειακά. Οφέλη ως προς την απασχόληση, την υγεία και την ασφάλεια. Ο στόχος αυτός, ήδη το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να λάβει υπόψη τη μείωση του κόστου των τεχνολογιών, είχε προτείνει ως πιο αποδοτικό ποσοστό μακροπρόθεσμα. Το είπε και στην ανταλλαγή απόψεων. Η ενέργεια και οι κλιματικές αλλαγές είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο συντονισμός των δράσεών μας για να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των στόχων μας και για, στο, και για την ενέργεια και για το κλίμα σε διαφορετικά επίπεδα, ε, η ευθυγράμμιση αυτή είναι απαραίτητη και θεωρώ ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση οδεύουμε προς το σωστό δρόμο. Ο κύριος Κάρινς τώρα, που είναι εισηγητής για το οικολογικό design. Ευχαριστώ. Ήδη οι συνάδελφοι έκαναν πολλά σχόλια. Θα επανέλθω σε κάτι που είπε στην αρχή ο Κλόντα Τούρμες. Ε, κάτι που άκουσα επανειλημμένος είναι μια έκκληση για ανάληψη δράσης προκειμένου να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Αναμφίβολα, αυτή είναι μια σημαντική πτυχή του θέματος. Κατά τη γνώμη μου και δεν νομίζω ότι είμαι μόνος ε, στην ομάδα μου, η Ενεργειακή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την πτυχή. Είναι κάτι πολύ πιο σφαιρικό. Και ακούγοντας τη συζήτηση, θυμήθηκα κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη μεταξύ των αγορών, πλήρης ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, ενεργειακή απόδοση, κλιματική δράση επίση και ε, ενέργεια, έρευνα, έρευνα μάλλον στην καινοδομή και τεχνολογική ανάπτυξη. Είναι πολλέ πτυχές ε, τη Ενεργειακή Ένωση. Είναι θέμα που βάζουμε την έμφαση και αν δεν θέσουμε τις αγορές στο επίκεντρο ε, γιατί η αγορά είναι ο βασικός πάροχος της ασφάλειας των επενδύσεων, που είναι ένα σημαντικός παράγοντας, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Οι αγορές ε, δεν ε, υπακούν σε ιδεολογίες, αλλά σε επενδύσεις. Χρειάζονται ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Θα πρέπει να αποδεσμευτούμε από τις επιδοτήσεις που στρέβλωνουν τις αγορές, είτε στα ορυκτά καύσιμα που έχουμε τέτοιες επενδύσεις, είτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αυτό συμβαίνει, αυτό συνέβη. Και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τα τελευταία πέντε χρόνια έγινε μια ε, τεχνολογική επανάσταση και οι τεχνολογίες για την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια είναι πια ανταγωνιστικές ε, με άλλες ε, παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως τα ορυκτά καύσιμα. Οπότε η ανάγκη να επιδοτήσουμε και τεχνητά να υποστηρίξουμε τις τεχνολογίες αυτές ε, θα, θα αποβεί βάρος των αγορών και ει βάρο των στόχων μας. Θέλουμε συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού. Έτσι θα προσελκύσουμε τις επενδύσεις. Και οι επενδύσεις ε, θα στραφούν και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί πια έχουν βελτιωθεί εκεί πολύ τα περιθώρια κέρδους και μακροπρόθεσμα επίσης. Και σίγουρα όλες οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες ε, ε, που πριν από πέντε χρόνια ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τα ρηκτά καύσιμα, θα διαπιστώσουν ότι και οι απέχουν λεφτά και θα... αλλά θα πρέπει να αποδεσμευτούμε, να απελευθερωθούμε από τις, επενδύσεις, από τις επιδοτήσεις. Οπότε δεν θα πρέπει να επικεντρώνουμε την Ενεργειακή Ένωση μόνο στις κλιματικές δράσεις. Ναι, δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα και σίγουρα θα ασχοληθούμε και με αυτό. Αλλά αν δεν κρατήσουμε τις, α... τις αγορές στο επίκεντρο, δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ούτε τους κλιματικούς μας στόχους. Οπότε δεν θα πρέπει να είμαστε μονομερείς εδώ. Και σίγουρα οι στόχοι μας ε, είναι πολύ πτυχοί και πολυεπίπεδοι. Αλλά αν δεν φέρουμε την αγορά στο επίκεντρο της προσπάθειας, δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε κανέναν από τους στόχους μας. Παρακαλώ, ρίχνετε και μια ματιά στο χρονόμετρο να αρχίσουν και να βοσβήνουν τα στεράκια, σημαίνει ότι τον έχετε υπερβεί. Ο κύριος Eckhout, που είναι συντάκτης γραμμοδότησης για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Από πλευρά ΕΝΒΗ, η οδηγία για τις ανανεώσιμες, αυτή με απασχολεί. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την διακυβέρνηση, γιατί εφόσον συζητάμε τις ανανεώσιμες, αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό είναι το επίπεδο φυσικά χρήσης, αλλά και πώς θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό θέλω να τονίσω. Όλοι συζητούν για την ε, ασφάλεια και τη βεβαιότητα για τους επενδυτές. Αλλά εάν θεωρούμε ότι εάν απλώς υπάρχει ε, αγορά, απλώς θα έρθουν οι επενδυτές, η διαφορά ε, είναι ότι έτσι είμαστε αφελείς. Το βασικό είναι να ξέρουν οι επενδυτές και ασφάλεια ε, οι επενδυτές λοιπόν να ξέρουν οι επενδυτές σε τι κατεύθυνση, κατεύθυνση θα πάει η Ευρώπη. Αυτό θέλουν οι επενδυτές. Υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις. Δεν υπάρχει επαρκής όμως σαφήνεια, βεβαιότητα. Πού θέλει να πάει η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Και μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές που έχουμε είναι η οδηγία μέχρι το 2020 για τι ανανεώσιμε, όχι μόνο για τους στόχους, αλλά γιατί έδωσε στα κράτη-μέλη μία κατεύθυνση να εργαστούν για να επιτύχουν ένα κάποιο επίπεδο. Αυτό λειτουργήσε. Έτσι κάναμε τη μετάβαση, την ξεκινήσαμε τουλάχιστον. Αυτό πρέπει να διατηρήσουμε και μετά το 2020. Αν εξετάσουμε το επίπεδο, είναι τρελό ότι τώρα που γίνονται ανταγωνιστικέ αυτέ τι τεχνολογίε και βλέπουμε τι αλλαγέ και μειώνεται ο βυθμό αύξηση. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αύξηση 5%. Μετά το 2020 η Επιτροπή προτείνει 1% ετήσια αύξηση. Αυτό είναι βλακώδες. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Και χαίρομαι που οι συγητές προτείνουν αυτή την αλλαγή και μαζί με τους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές για το θέμα των ανανοσίμων θα κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάουτ. Ρόιντα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ρόιλ. Ρόιλ. Να ασχοληθώ με δύο θέματα. να μου πει γραμματεία τις επόμενες μέρες αν είναι σωστό ότι τώρα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό της η διακυβέρνηση και έτσι στην ουσία ασχολούμεθα ιδιαίτερα με αυτήν ενώ έχουμε πολλά άλλα. Δεν καταλαβαίνω. Συζητάμε ε, ε, θέματα τα οποία θα διευκρινιστούν σε άλλες οδηγίες. Είναι δυνατόν να αλλάξει τόσο πολύ το κείμενο της Κομισιόν η διακυβέρνηση να γίνει ένα πολιτικό πρόγραμμα που στην ουσία αποτελεί το πλαίσιο για όλες τις άλλες πολιτικές. Είναι δυνατό, είναι κατανοητό κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να το καταλάβω γιατί αλλιώ μπορούμε να σταματήσουμε την ε, εργασία για τα άλλα θέματα. Αν ξεκινήσουμε με ένα θέμα που ούτως ή άλλως αδειάζει με περιεχόμενο όλα τα άλλα. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω, αν επιτρέπετε, να, πάμε, να πηγαίνουμε τόσο βαθιά. Αναφέρθηκε ένα σημείο. Ελαστικότητα, ευελιξία, ο ρόλος των κρατών μελών για το ενεργειακό μείγμα. Δεν είναι δυνατόν να τα λύσουμε αυτά τα θέματα με μια νομική ρύθμιση. Δεν έχει καμία έννοια να αντιμετωπίζουμε έτσι το θέμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η διακυβέρνηση ε, τίθεται με τόση τρομερή προτεραιότητα. Μπορούμε βεβαίω να εργαστούμε με το κείμενο τη Κομισιόν να το αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε εντελώ να το ανατρέψουμε. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Η κυρία ε, Φαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά υπόθηκαν. Πολύ ενδιαφέρον που είμαστε μαζί συνάδελφοι Ένβη ε, και Ήτρε. Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομη. Έχω δύο λεπτά. Πολιτικό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να πω. Βεβαίως το πακέτο της καθαρής ενέργειας έχει πολλούς στόχους. Αλλά για την πολιτική μας ομάδα ο βασικός στόχος είναι η εφαρμογή της συμφωνίας COP21. Βλέπετε τι ζέστη έχει σήμερα. Και μπορεί να μας αρέσει η ζέστη. Αλλά βγήκε μια νέα έκθεση που λέει ότι οι καύσονες θα γίνουν πολύ επικίνδυνοι στο μέλλον. Όχι μόνο σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά και στην Ευρώπη. Άρα η εφαρμογή της συμφωνίας COP21 είναι βασικό σημείο για την καθαρή ενέργεια. Δεύτερον, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια είναι πακέτο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί αυτή η ολιστική αντιμετώπιση. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν αντιφάσει ανάμεσα στα μέρη. Γι' αυτό είναι θέμα κλειδί η διακυβέρνηση. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο. Συντονίζει τα διάφορα επιμέρους. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε αυτό πάντα υπόψη μας. Το βασικό δεν είναι το α ή το β τμήμα, αλλά η διακυβέρνηση. Οπότε, οπότε είναι πολύ καλή η αρχική προσέγγιση των εισηγητών. Πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη θεώρηση. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το 2050 και με βάση το 2050 να καθορίσουμε μετά τα νωρίτερα. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Στρατηγική, ολιστική προσέγγιση. Είναι νέα προσέγγιση, αλλά θεωρώ ότι είναι απόλυτα αναγκαία να υπάρχει η σωστή, ο σωστός καταμερισμός μεταξύ αυτών που αποφασίζουμε στις Βρυξέλλες και αυτών που εφαρμόζονται στην πράξη, στις περιφέρειες, στην πολιτική, γιατί εκεί εφαρμόζεται η κλιματική πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Λίζε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση ΙΤΡΑ και ΕΝΒΗ, γιατί έχω εργαστεί και για τις δύο επιτροπές, τώρα είμαι μόνο στην ΕΝΒΗ και νομίζω ότι είναι βλακώδες να ε, αντικρούμε ο ένας τον άλλον. Αντίθετα, πρέπει να συνεργαζόμεθα. Ως Επιτροπή Ένβη θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι των Παρισίων. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάπως πιο συγκεκριμένες τις διατυπώσεις. Πιο σαφείς και να δούμε πως είναι και υπερβολικά φιλόδοξοι κάποιοι. Στο Παρίσι ε, αναφέρεται ο στόχος 1,5 ε, βαθμός, αλλά και 2 βαθμοί, να είμαστε δηλαδή στο 80-95% της ανώτερης ε, λωρίδας της ε, κλίμακας, βεβαίω είναι πολύ σημαντικό η τεχνολογία να είναι ουδέτερη. Γι' αυτό εκτιμώ τις ε, ε ανανεώσιμες και τις ε, προωθώ. Αλλά αν το 2050 δεν θα έχουμε και άλλες τεχνολογίες που δεν μπορούμε σήμερα να τις προβλέψουμε. Μήπως θέλεις, λέει ο κύριος Τούρμες, και πυρηνική ενέργεια για τη Γερμανία. Όχι, δεν θέλω πυρηνική ενέργεια για τη Γερμανία, λέει ο κύριος Λίζε, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπου θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση. Η στόχη το 2030 πρέπει να καθοριστούν σαφώς και να περιγράψουμε και πώς θα τους επιτύχουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στόχημη εθνικά δεσμευτική. Δεν είναι, συγγνώμη, σκόπιμη εθνικά δεσμευτική στόχη. Να μιλήσουμε με, για άλλα ορόσημα για να μην τιμωρηθούν όσοι κάνουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια αν δεν επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι συνολικά. Επίσης πρέπει να είμαστε ρεαλιστές το 5% κλόν δεν νομίζω ότι το λέω σοβαρά. Η θέση του Κοινοβουλίου από το 14 και είναι η θέση η Τρένβη που λέει 30%. Συγγνώμη, το 45% ε, είναι υπερβολικό. Πρέπει να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και μετά να συζητάμε και για το πώς θα τους επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ελίζα. Η κυρία Ντελκαστήλιο Βέρα. χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ε, θα είμαι λακωνική και δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα των προλαλισσάντων, ε, κυρίως των συναδέλφων της πολιτικής μου ομάδας από την Ήτρε. Θα ήθελα να μιλήσω για τους μηχανισμούς, για τα εργαλεία μας, γιατί χρειαζόμαστε εργαλεία για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Μηχανισμούς και εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες ε, των διαφόρων χωρών, γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και διαφορά στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτή την άποψη οι διασυνδέσεις θα έχουν ευραλγικό ρόλο από πολλές και διάφορες απόψεις. Θα έχουν κέριο ρόλο για την ασφάλεια, την ενεργειακή, για την ε, αγορά της Ενεργειακής Ένωσης και για την υλοποίηση των στόχων που θα θεσπίσουμε και για το κλίμα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε εργαλεία και θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να ε, φροντίσουμε να δώσουμε σάρκα και οστά στο στόχο της διασύνδεσης. Γιατί έτσι θα μπορέσουν και κράτη-μέλη που υστερούν να υλοποιήσουν τους στόχους για το 2020 και φυσικά για το 2030 που στόχο έχουμε το 50% για τις διασυνδέσεις. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις γιατί θα είναι κέριος επαναλαμβάνω ο ρόλος τους και κυρίως ε, για χώρες ε, όπως η Ιρλανδία, η Πολωνία και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανανάτο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη υπόθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ παίρνω το λόγο για να εκφράσω την γενική μου υποστήριξη στο σχέδιο έκθεσης που παρουσίασαν οι συνάδελφοί Τούρμες και Ριβαζή. Βεβαίω, ε, συμμερίζομαι ιδιαίτερα την ανάγκη ευθυγράμμιση του στόχων ε, κλίματος και ενέργειας ε, για το, ε, ορίζοντα το 2030 με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στη Παρίσι εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση. Ωστόσο πρέπει να τονίσω ότι η αναθεώρηση τονίζει το στόχο για τις ανανεώσιμες, σε πράγμα το οποίο τόνισαν οι πράσινοι, αλλά παρουσιάζει κάποια προβλήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις και όχι το σημείο άφεξης. Ε, είμαστε λοιπόν μέσα σε ένα διαθεσμικό θέσιο που θα καλύψει πολλά θέματα ταυτόχρονα και είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους. Θεωρούμε ότι οι στόχοι που αναφέρονται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση θα πρέπει να συντονιστούν με τις ε, τομεακές νομοθεσίες ε, ε, όπως αυτήν για τις οποίες εργάζεται ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Και άρα θα πρέπει να βρεθούν συμβιβαστικές τις οποίες να στηρίζει μια μεγάλη πλειοψηφία. Να το υπογραμμίσω επίσης και εδώ συμφωνώ πολύ με τη συνάδελφο Γκρίφιν και τον συνάδελφο Ζωρίνιο εδώ δίπλα μου ότι χρειάζεται δηλαδή να εκπονήσουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με αφιερωμένη στους εργαζόμενους και τις ε, τοπικές ε, ε, αρχές ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης από την ενεργειακή μετάβαση έτσι ώστε να ευνοηθούν οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε καθαρές τεχνολογίες και αυτό στις κοινότητες που περισσότερο από όλες θα υπέφεραν λόγω της ε, πάυσης χρήσης του άνθρακα. Αυτά με βάση τις συστάσεις της Επιτροπής, ώστε να δεσμευτούμε ε, αλλά χωρίς να επιβαρύνουμε περισσότερο τους, τους φορείς και να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη κατανομή της προσπάθειας αυτής και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ και τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κόχλιτσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμπρός, με ακούτε?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 Σας ευχαριστώ. Κάτσε στη θέση άλλου, άλλης μάλλον. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τα θέματα αυτά, αλλά από πολιτική άποψη, όχι από τεχνική. Είναι καλό ότι έχουμε μια πολιτική απόφαση και έχουμε και στόχους, τους στόχους του Παρισιού, αλλά η πολιτική συζήτηση χωρίς τεχνικό υπόβαθρο είναι ε, απαράδεκτη ή μάλλον ανέφικτη η ε, υλοποίηση των στόχων μας αν δεν έχουμε πρώτα κάποια τεχνικά θεμέλια. Ε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τρευλώνουν την ενεργειακή αγορά και δεν δίνουν καμία πραγματική όθηση. Και οι Γερμανοί είναι καλό παράδειγμα στρέβλωσης ε, της αγοράς που δεν δίνει ενάυσματα για την αλλαγή των ρυθμίσεων. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις για το πακέτο. Κάποιος αναφέρθηκε στο μεθάνιο, στις εκπομπές μεθανίου που είναι πολύ πιο επιζήμιες για το περιβάλλον ε, από ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και παρόλα αυτά δεν λέμε τίποτα για το μεθάνιο το παραβλέπουμε πλήρως. Επίσης, ε, τα φωτοβολταϊκά και η αιωλική ενέργεια θα μπορούσαν να, να ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να έχουμε επαρκείς πόρους. ένα τρίτο του χρόνου έχουμε αέρα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ ε, στη, στη Βόρεια Ευρώπη έχουμε 70% του χρόνου να φυσάει ο αέρας. Και τι γίνεται τον υπόλοιπο χρόνο. Θα σταματήσει η βιολογική παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το πακέτο, γιατί μερικές φορές ε, μιλάμε σαν να μην έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, με πεδαριώδη τρόπο. Θα πρέπει να προβλέψουμε πρώτα τεχνικές λύσεις. Οι Γερμανοί μας απέδειξαν ότι είναι δυνατόν να κρατήσουμε και ορυκτά καύσιμα και χρυσή άνθρακα για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε συμπερίληψη στο δίκτυο όλων των διάφορων μορφών ενέργειας και γι αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Αγιούσο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω λίγα πράγματα. Καλή και άγιοι στόχοι αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύουμε ηλεκτρισμό όπως το κάνουμε με το νερό. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε 15% στόχο για τις διασυνδέσεις. Το 2000-2001 προτάθηκε το 10% και είδατε που βρεθήκαμε σήμερα. Ε, και δεσμευτική είναι η στόχη, αν δεν πληρούνται μπορούμε να το λέμε στα χαρτιά, αλλά δεν θα δημιουργήσουμε ποτέ μια γνήσια ενεργειακή αγορά. Ούτε πρόκειται να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους γιατί η παραγόμενη ενέργεια θα μπορέσουμε να τη, την παραγόμενη ενέργεια θα μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε από το ένα σημείο στο άλλο δυστυχώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώτα η κυρια κυρία Ρίτσαρτς. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω, ε, πολύ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συζητώ μαζί σας αυτή την πρόταση, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό ε, στοιχείο του πακέτου για, την, ε, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την καθαρή ενέργεια. Πολλοί ε, μίλησαν για την ανάγκη επιδίωξης των στόχων του Παρισιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ε, έχουμε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής και έρχομαι εδώ με τους συναδέλφους και από την Επιτροπή, από την Διεύθυνση για το Περιβάλλον. Θέλουμε φυσικά ε, καθαρότερη ενέργεια, αποδοτικότερη ενέργεια, θέλουμε αύξηση της απασχόλησης των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόθεση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο. Γι' αυτό και το πακέτο της διακυβέρνησης είναι τόσο σημαντικό γιατί συγκενά αυτά τα στοιχεία, τα συνδυάζει και μας επιτρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση και περιμένω και την έκθεση μετά τα σχόλια του εισηγητού. Κατά τη γνώμη μας, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι να κρατήσουμε αμύωτο το επίπεδο φιλοδοξίας ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι σημαντικό, να παραμείνουν υψηλές οι φιλοδοξίες μας ε, και σε ό,τι αφορά τους δεσμευτικούς στόχους για τα εθνικά σχέδια, ε, τη, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τα μέτρα σε περίπτωση που έχουμε μια υστέρηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους. Και φυσικά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να ενισχύσουμε τις ε, διατάξεις και να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για την Ενεργειακή Ένωση και για το κλίμα για το 2030 και να τηρήσουμε και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Και χάρη στο πακέτο αυτό θα υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους που συλλογικά έχουμε αναλάβει. Και όπως είπα και οι Πρόεδροι επανειλημμένος, είναι σημαντικό αυτό το πακέτο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον ακέραιο χαρακτήρα του. Έχουμε 8 νομοθετικές πράξεις που προτείνονται με στόχους ε, σε τομεακές νομοθετικές προτάσεις. Θα πρέπει όμως να διαφυλάξουμε αυτή την σφαιρική αλληλεπίδραση και την σύνδεση των τμήματων, τα οποία είναι αναπόσπαστα στο συνολικό πακέτο. Και επαναλαμβάνω, η σφαιρική προσέγγιση, η ολιστική προσέγγιση είναι σημαντικό. Ε, και στην καθαρή ενέργεια θα πρέπει να μείνουμε στους στόχους του 2030 και να μην μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εθνικές γραμμικές πορείες, κάτι που θα μας επιτρέπει να θα μας επιτρέψει να αποτιμήσουμε την εθνική πρόοδο σε ένα χρονικό ορίζοντα. Και φυσικά και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο αυτό θα είναι σημαντικός. Κάτι άλλο που είπα προηγουμένως είναι η ανάγκη σφαιρικής προσέγγισης, ολιστικής προσέγγισης. Το λέω και θα το επαναλάβω. Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν και τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Φυσικά, επίσης, η ιδέα... Ε, σχεδίων και προγραμμάτων ενεργειακού ενδιαφέροντος ευρωπαϊκού είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε πιο διεξοδικά άλλη στιγμή. Θα πρέπει να συνδέσουμε τις επενδύσεις με την ανταγωνιστικότητα, όπως είπατε και είναι πολύ σημαντικό θέμα, να ενθαρρύνουμε ιδιώτες επενδυτές να επενδύσουν στους κλάδους αυτούς. Ήδη βλέπουμε ρηξικέλευτες αλλαγές ε, τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό και είμαι πεπισμένη ότι ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση θα προωθήσει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα που χρειάζονται οι επενδυτές και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας στον ενεργειακό κλάδο. Κάτι άλλο. Η δυνατότητα του άρθρου 14 για την αναβάθμιση της φιλοδοξίας των σχεδίων. Αναβάθμιση όμως μόνο, όχι υποβάθμιση. Η αναθεώρηση των φιλοδοξιών μόνο προς τα πάνω γίνεται και όχι για μείωσή τους. Επίσης, είμαστε υπέρ μιας ισχυρής περιφερειακής συνεργασίας που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα περιφερειακά στοιχεία διασύνδεσης και συνεργασίας εξαρτώνται από τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη ανάμειξη των ενδιαφερομένων, όπως είπατε. Ήταν σαφές και από τη συζήτηση και για μας είναι πολύ σημαντικό. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για να έχουμε απαραίτητη δημοκρατική ε, συμμετοχή και έλεγχο. Επίσης, το θέμα της ενεργειακής φτώχειας, ο λόγος των, ε, των πολιτών, διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, την κοινωνία των πολιτών, απασχόληση, ανάπτυξη, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, θέλουμε φιλόδοξα εθνικά σχέδια θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και φυσικά σημαντικός ο ρόλος των ευρωπαϊκών και των εθνικών εταίρων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στην πορεία. Επαναλαμβάνω, θα κρατήσουμε αμύωτη την πίεση για να επισπεύσουμε τα πράγματα και να διεκπαιρέσουμε το πακέτο το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέκμαν από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Και εσείς παρακαλώ δύο-τρία λεπτά, όχι παραπάνω. Ναι, βεβαίως θα προσπαθήσω. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ε, ε, ολοκλήρωση κλίματος και ενέργειας όπως τη βλέπουμε στην πρόταση, το βλέπουμε και από τις παρεμβάσεις εδώ, αλλά το βλέπουμε και ευρύτερα στην κοινωνία αλλά φυσικά και την εφαρμογή των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι περιλαμβάνονται πολλές καλές ιδέες στην πρόταση ε, διακυβέρνησης που είναι ήδη φιλόδοξη από μόνη της. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια κοινή πρόταση για την ενέργεια και το κλίμα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτά τα βασικά στοιχεία όπως έχουν και να τα συζητήσουμε. Κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και βεβαίως έχουμε ακούσει για μακροπρόθεσμες στατικικές που ακολουθούν τα σχέδια μπορεί να είναι με αυτό παράλογο, αλλά είδαμε ότι, ανάγκη να έχουμε, ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε τη, τα σχέδια νωρίτερα γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε το Παρίσι, ενώ οι δομές παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο και θα πρέπει να είναι αυτά τα δύο συμβατά μεταξύ τους και έχουμε χρόνο να το επεξεργαστούμε ώστε μακροπρόθεσμα αυτά τα σχέδια και οι στρατηγικές να είναι συνεπεί μεταξύ τους και να αλληλοϊποστηρίζονται. Και βεβαίως έχουμε και την ενημέρωση των σχεδίων κάθε πέντε χρόνια που μπορούν, μπορεί να λάβει υπόψη τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Να πω επίσης σε αυτό το πλαίσιο από το σχέδιο έκθεσης ότι έχουμε πολύ καλές ιδέες και οι κλιματικέ αλλαγές όντως πρέπει να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Τώρα για το 2050 νομίζω πως είναι κάπως νωρί, γιατί η δουλειά τώρα θα αρχίσει στα κρατημέλη και στην Επιτροπή επί τη βάση των δύο αξιολογήσεων καθώς και των διαβουλεύσεων με τους ε, ε, φορείς και την αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτό σε σχέση με τον 1,5 βαθμό, το στόχο του 1,5 βαθμού, είναι σημαντικό, δεν ξέρουμε κατά πόσο η επίσης θα καλύψει αυτή την έκθεση. Ίσως θα πρέπει εκεί να περιμένουμε για να, πριν λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις. Ενδιάμεση στρατηγική, η, μεσο, η μεσο Η στρατηγική για το μεθάνιο ε, έχουμε δουλέψει πολύ και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές, αλλά Ίσως να μην είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε ολόκληρη στρατηγική σε αυτή τη φάση και να πω και δύο λόγια για το ETS. Το ETS έχει το ίδιο το δικό του σύστημα διακυβέρνησης, είναι ένα οικονομικό ε, μέσο και γι' αυτό και προτείνουμε να μην επαναλάβουμε κάτι που ήδη υπόρχει. Υπάρχει πάντως συντονισμός ανάμεσα στο ETS και την διακυβέρνηση. Νομίζω πως αυτά είχα να πω τρία λεπτά. Και αν μην είχατε μιλήσει πέντε λεπτά θα ήταν βέβαια περισσότερο εισόδημα, αλλά κύριε Τούρμες, θα δώσω την ε, άλλη φορά το λόγο στον κύριο, μόνο στην κυρία Ριβαζή. Θα ήθελα να δώσω μια πιο αναλυτική απάντηση. Αλλά πολλοί συνάδελφοι βαίνεται ότι πεινούσαν. Θα είμαι σύντομος. Σήμερα μου έκανε το, τη μεγαλύτερη φιλοφρόνηση που θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ένας συνάδελφος του ΕΛΚ. Κρίμα που έφυγε ο Χέρμπερτ. Γιατί είπε ακριβώς αυτό που θέλω και πρέπει να κάνω. Η διακυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα, όπως είπε, Gesamtkunstwerk, δηλαδή ένα συνολικό οικοδόμημα, ένα συνολικό έργο τέχνης για να επιτύχουμε το Παρίσι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο αν κινητοποιήσουμε εκατομμύρια πολιτών. Ναι, είναι Gesamtkunstwerk και ελπίζω να το επιτύχουμε. Ο κύριος Κάρενς είπε ότι ασχολούμεθα πολύ με την ε, κλιματική αλλαγή. Ξέρετε ο, ποιος μας έκανε τη μεγαλύτερη φιλοφρόνηση για την ε, κλιματική μας πολιτική και την περιβαλλοντική μας πολιτική τις τελευταίες 15 ετίες. Ο Πούτιν που δημοσίευσε ένα κείμενο για την οικονομική πολιτική και την πολιτική ασφάλιση και κάνει μια παράγραφο που λέει, περιέχει μια παράγραφο που λέει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη ρωσική οικονομία είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα της Ευρώπης και οι πράσινες τεχνολογίες. ο κύριος Πούτιν επιτέλους κατάλαβε ότι αυτό που κάνουμε αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα. Για μας το μεγαλύτερο θέμα ενεργειακής ασφάλειας είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση ακόμη περισσότερο και να περάσουμε ακόμη ταχύτερα στις ανανεώσιμες. Έτσι θα έχουμε ασφάλεια, όχι μόνο για την ενέργεια. Αυτό μας φέρνει και γεωπολιτική ασφάλεια. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τώρα είμαστε εμείς, η Ινδία και η Κίνα, που είμαστε στην πρωτοπορία της τεχνολογικής αλλαγής, κερδίζουμε τη μάχη έναντι εκείνων που είχαν τεράστια αποθέματα πετρελαίου, το οποίο δεν αξίζει πια 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν αξίζει, η τιμή του δεν είναι ούτε καν 50 ή 40 δολάρια. Γιατί? Γιατί ήμασταν τόσο καταπληκτικοί τα τελευταία χρόνια που αλλάζουμε προς όφελός μας τη γεωπολιτική κατάσταση. Για τις αγορές κρίμα που έφυγε ο κύριο Κάριν, Αγαπητοί Ισπανοί συνάδελφοι, αν θέλετε να υπάρχει διασύνδεση Γαλλίας και Ισπανίας, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα σας το παράσχουν οι αγορές. Αν ο κύριος Κάρενς θέλει μια πλήρη οικονομία της αγοράς να πει στους Ισπανούς συναδέλφους να μην υπάρχει αγωγός από τη Γαλλία στη Γερμανία. Και αν δεν υπάρχει αυτή η αγορός, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα είναι τρομερά φτηνά Πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ε, καινοτομία στην Ευρώπη, ή μάλλον την ε, συντήρηση και ανακαίνιση της υποδομής. Θα χρειαστούν δημόσιες υποδομές. Θα χρειαστούμε και δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων με πολύ υψηλού επίπεδου σχεδιασμένη θεσμική πλαισίωση, θεσμικό πλαίσιο. Και το θετικό είναι ότι έχουμε 3 εκατομμύρια από τα συνταξιδοτικά ταμεία που σπρώχνονται για να επενδύσουν. Να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες για απόδοση 3, 4, 5%. Τέλος. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Νομίζω ότι εμείς είμαστε στο τιμόνι της προσπάθειας και λυπάμαι για την Γενική Διεύθυνση για το κλίμα. Σας παρακαλώ αυτά που έχετε επιτύχει τα τελευταία δέκα χρόνια. Σκεφτείτε δηλαδή, το ETS, γιατί πρέπει να σας απασχολεί μόνο αυτό. Λέτε ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο φιλόδοξοι για το 2050. Ας είμαστε χαλαροί. Σας παρακαλώ, ξαναδείτε τα δεδομένα σας. Ο κύριος ε, Κανιέτε είναι πιο προευτικός σήμερα από εσά και τον κύριο Τελμπέκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτική τελικά ε, είναι επικεφαλής. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που είπατε σήμερα το πρωί, για τόσα θέματα, για να συνδυαστεί το 2050 και το 2030, για να είμαστε φιλόδοξοι. Ξέρετε ότι βρέχει στην Αντρακτική. Καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Δεν είχε βρέξει ποτέ. Αρχίζει να βρέχει στην Ανταρκτική, τότε είμαστε πολύ κοντά στο σημείο καμπή. Και θα συνεχίσει να βρέχει στην Ανταρκτική. Θα λιώσει ο πάγο. Και δεν θέλω γενική, οι δημόσιοι πάλι από τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος να μου λένε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο ε, Κλοντ, λέει ο πρόεδρος, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Έχουμε κάποιους κανόνες, ε, ξέρετε, ευγένεια και θέλουμε να τηρήσουμε και το χρόνο μας. Είχατε πολύ χρόνο για να μιλήσετε. Με συγχωρείτε, πρέπει να σας διακόψω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι έχεις επιτύχει. Και σε συγχαίρουμε. Αντίνα. Ευχαριστώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Εκτός αν θέλει να πει τίποτα η Γενική Διεύθυνση για το κλίματος, επειδή υπέστη επίθεση. Αλλά δεν αφορούσε βέβαια η επίθεση προσωπικά τον κύριο Μπέγκμαν. Θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Αν έτσι ερμήνευσε ο κύριο Τούρμες αυτό που είπε, λυπάμαι γι' αυτό. Η Γενική Διεύθυνση Κλίματος οπωσδήποτε αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά σοβαρότερα από οποιονδήποτε άλλο. Έχουμε το ETS, ε το έχουμε DSR, έχουμε το LULUSF, όλα αυτά επίκεντρα, έχουμε το 2050. Εργαζόμαστε πολύ γι' αυτό. Εργαζόμαστε πολύ για να κάνουμε την στρατηγική μας για, για τα μέσα του αιώνα ακόμη πιο φιλόδοξη. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαζόμεθα, συγγνώμη, να εργαζόμεθα με το σωστό τρόπο. Αλλά βέβαια δεν λέω ότι πρέπει να επιβραδύνουμε. Συμφωνώ ότι αυτά που, που γίνονται τώρα και νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Άρια Κανιέτε, αυτό που κάνει ο Τραμπ μας κάνει ακόμη πιο ε, αποφασισμένους να, να κινηθούμε ταχύτερα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ε, εκπροσωπώ επισήμως την Ήτρε, πρέπει να σας πω αγαπητοί φίλοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν συμμερίζονται όλοι στην Ήτρε αυτά που είπε ακριβώς ο κύριος ε, Τούρμες. Πρέπει νομίζω ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς όταν μιλάμε. Θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους από την Ήτρε ελπίζω να μην χάσατε όλη σας την ενέργεια γιατί στις 3 η ώρα Έχουμε την επόμενη συνεδρίαση. όπου θα συναντηθούμε με όλους του επιτρόπους με τους οποίους εργαζόμαστε για την έρευνα, για την εσωτερική αγορά κλπ. Λοιπόν, έχουμε τρεις σημαντικές συζητήσεις με τους επιτρόπους μας. Αρχίζουμε στις τρεις. Σας παρακαλώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το... Committee e chair. You can finish our meeting Μπορείτε να ολοκληρώσετε την συνεδρίασή μας. Η προθεσμία για τις, ε, για τροπολογίες είναι ε, η 27 το μεσημέρι του μήνα. Και η συζήτηση θα γίνει στις 11 Ιουλίου από 19 το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπούζακ. ευχαριστώ πολύ πολύ φορά.